Εντάξει. Το οριστικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης ε, εγκρίθηκε στις 6 Δεκεμβρίου από τη διάσκεψη των ε, Προέδρων και έχει διανεμηθεί. Έχει καθοριστεί λοιπόν έτσι η διάταξη των εργασιών. Ας προχωρήσουμε λοιπόν με την ημερήσια διάταξη που προβλέπει την ε, συζήτηση